Μαρίου είναι η προθεσμία για τροπολογίες και Τετάρτη έχουμε την ε, ψηφοφορία από τις αρμόδιες αρχές της Δανίας. Ε, πληροφορηθήκαμε πως εξελέγει ο κύριος Κλάους Λάρσεν Γένσεν, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Γιώργενσεν με ισχύ από τις 13 Δεκεμβρίου 2013. Ο κύριος Γιώργενσεν έγινε υπουργό. Οι αρμόδιες αρχές Πολωνίας με ενημέρωσαν για την ε, εκλογή δύο συναδέλφων, ο κύριος Μπιγνιέφ Ζαλέσκη, ο οποίος αδικαστητά την κυρία Κολάρσκα Μπομπίντσκα και ο κύριος ε, Ταντέος Ρόστιτ, ο οποίος αντικαθιστά τον κύριο Ραφάλ Τσασκόφσκι. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 4